την αξιολόγηση αντικτύπου ο Αντιπρόεδρος Τσίμερμαν να θα λάβει το λόγο μόλις καθίσει για να κάνει τη δήλωση αυτή. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Επιτρέψτε μου να πω πόσο σημαντική είναι η αξιολόγηση αντικτύπου για αυτή την Επιτροπή. Θα πρέπει να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη, την απασχόληση, να μην επιβαρύνουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με άσκοπη νομοθεσία. Πρέπει να προβλέψουμε ώστε να παραδίδουμε τα απαραίτητα και αναγκαία για να ε, βεβαιωθούμε ότι θα αξιοποιήσουμε τις ε, δυνατότητες της οικονομίας που μένουν αξιοποιείται σήμερα. Πιστεύουμε ότι οι τρει μα θεσμικά όργανα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ευθύνη να αξιολογούν κατά, την, κατά το, τη διαδικασία του νομοθετή ότι η νομοθεσία επιτυγχάνει του στόχου, τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Γι' αυτό είμαι πεπισμένος στην αξιολο... Ε, για την ανάγκη της αξιολόγησης αντικτύπου όταν προετοιμάζεται το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρειάζονται βελτιώσεις και στο πώς γίνεται η αξιολόγηση αντικτύπου από την Επιτροπή και πώς το Συμβούλιο Αξιολόγησης Αντικτύπου ε, θα μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Πιστεύω κύριε Πρόεδρε ότι έχουμε κοινή ευθύνη με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν μου επιτρέπετε, για να βελτιώσουμε την αξιολόγηση αντικτύπου στην πορεία. Γιατί σε τελευταία ανάλυση αυτό που έχει αντίκτυπο δεν είναι η πρόταση όπως αρχίζει στη νομοθετική διαδικασία, αλλά η έκβαση ε, τη νομοθετική διαδικασία είναι σημαντική και όλοι γνωρίζουμε ότι δεν μιλάμε κατά ανάγκη για τα ίδια πράγματα. Αυτό που χρειάζεται εννοώ είναι να βελτιώσουμε Ξέρω ότι συμφωνείτε. Θέλουμε λοιπόν να φροντίσουμε ώστε παράλληλα με τις διαδικασίες να γίνεται αξιολόγηση αντικτύπου από τα τρία θεσμικά όργανα. Όταν δηλαδή αποφαινόμεθα για μια οδηγία και πριν αυτή περάσει και ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία να φροντίσουμε να βεβαιωθούμε ότι θα γνωρίζουμε καλά τον αντίκτυπο αυτής της οδηγίας, του τι αποφασίζουμε να κάνουμε και πώς θα φροντίσουμε ώστε αυτό που θα κάνει θα ε, αποσκοπεί στο στόχο που έχουμε θέσει, τίποτε περισσότερο. Όπως είπα στην ακρόαση, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, όλος ιδιαίτερα, να βοηθήσω με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που έχουν. Σε διάφορες μελέτες που γνωρίζω και από τις επαφές που έκανα με αρχές αξιολόγησης αντικτύπου στα κράτη-μέλη, ε, μου έγινε σαφές ότι η απάλληψη κάποιων διοικητικών εμποδίων ή άσκοπων ρυθμίσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να παίξει καταλητικό ρόλο στην καταπολέμηση της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φανταστείτε για να κάνουμε συζήτηση. Θεωρητικά ότι μπορούμε να άρωμε την, το διοικητικό ε, φόρτο κατά 10% ενός επαγγελματία ενός κρεοπόλη, ενός αρτοπιού. Αυτό μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή μπορεί να επιτρέψουν στον κρεοπόλη, στον αρτοπιό να προσλάβουν έναν ακόμα. Ή από την άλλη, το χειρότερο σενάριο, ε, να τον αναγκάσουμε να κλείσει την επιχείρηση. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα μπορεί να δώσουν πάρα πολύ μεγάλα αποτελέσματα γιατί δεδομένου του, του αριθμού των ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν τις βοηθήσουμε, θα βοηθήσουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση. Σας υπενθυμίζω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 85% των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα είναι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν λοιπόν βοηθήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις, έροντας κάποιο από το διοικητικό φόρτο, φροντίζοντας ότι όταν νομοθετούμε για αυτές θα ε, ε, αποσκοπούμε στην επίτευξη του στόχου μας ακριβώς αυτό είναι άμεση συμβολή στη δημιουργία μεγαλύτερης απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είμαι προσιλωμένος στο στόχο αυτό, είμαι έτοιμος να έλθω και να λογοδοτήσω σε εσά σε σχέση με αυτό το στόχο. Όμως χρειάζομαι απελπισμένο θα έλεγα την υποστήριξή σας, γιατί όταν αναλαμβάνει η δράση το Κοινοβούλιο στα πλαίσια της αξιολόγησης αντικτύπου, ε, ε, ε, η συμβολή του είναι πολύ μεγάλη. Δεν μπορούμε μόνοι μας ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το χρειαζόμαστε το Κοινοβούλιο και από το Κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα πείσουν το Συμβούλιο να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, γιατί μέχρι τώρα το Συμβούλιο δεν ήταν πολύ δραστήριο για να το πω ήπια ε, δεν ακολούθησαν δηλαδή ε, τα δύο άλλα θεσμικά όργανα στην επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη δήλωση αυτή. Και τώρα προχωρούμε στους ε, μιλητές από τις πολιτικές ομάδες. Ο συνάδελφος Μάρκους Πίπερ είναι ο πρώτος ομιλητής από την πλευρά του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ με τα μεσαία στρώματα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοβαλιά της ε, ε, οικονομίας και δεν πρέπει να πνίγονται από τη γραφειοκρατία. Στους πολιτικούς λόγους μας το λέμε αυτό και ο δικός σας λόγος ε, ήταν τέτοιος παρόλο που έχει και ουσία και προσανατολίζεται στο μέλλον. Καλέσατε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βοηθήσει και να αρχίσει το έργο αυτό από σήμερα ήδη. Θέλω να σας κάνω λοιπόν κάποιες ερωτήσεις ιδιαίτερα εις ό,τι αφορά τις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση αντικτύπου της Επιτροπής. Γιατί δεν υπάρχει πλέον ε, υποχρεωτική εξέταση των ε, ΜΜΕ γιατί ε, οι υπηρεσίες δεν είναι σαφώς προσδιορισμένες ως προς τα καθήκοντα, γιατί οι γενικοί διευθυντές πήραν μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια για το αν θα υπάρξει ε, εξολόγηση αντικτύπου ή όχι. Πρόκειται για πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις, αλλά θέλουμε να καλέσουμε την Κομισιόν, παρακαλώ, αυτό το τεστ των ΜΜΕ να το καταστήσουν πάλι υποχρεωτικό και να πάρουν πολύ στα σοβαρά τον αντίκτυπο, την αξιολόγηση αντικτύπου. Ε, ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε την πρωτοβουλία μας και ανεξάρτητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για, έχουμε στη Σουηδία, την Τσεχία, τη Μεγάλη Βρετανία και στη Γερμανία αξιολογούν ανεξάρτητη φορείς την αρμοδιότητα και τις γραφειοκρατικές επιπτώσεις της εθνικής νομοθεσίας. Γιατί να μην γίνεται αυτό και σε επίπεδο Βρυξελών. Μία ε, ε, ε, ανεξάρτητη αξιολόγηση αντικτύπου. Δεν θα πρέπει βέβαια να υποκαταστήσει κανείς το, το έργο της Κομισιόν ούτε το δικαίωμα ανάληψη πρωτοβουλία. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν μολόχο υπηρεσιών. Θέλουμε όμω να υπάρχει δυνατότητα διαβούλευση στα πλαίσια τη επικουρικότητα. Θα πρέπει να αποδείξουμε στους πολίτες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ομοθεσία της δεν χάνει το στόχο. Η ανεξαρτησία και η ε, αξιοπιστία μας θα βελτιωθεί. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τους ομιλητές μην, μην ξεπερνάτε τα χρονικά όρια. Ε, ευχαριστώ πολύ, Κρέσκο. Ένα λεπτό. Σοσιαλδημοκράτες. Αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε μια πραγματική δημόσια πολιτική. Γι' αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε αυτή τη συλλογιστική και να δούμε πώς μπορούν να πραγματοθούν όλα αυτά. Πιστεύω ότι αυτή η αξιολόγηση αντικτύπου έχει σημασία για να έχουμε ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες, έτσι ώστε να ξέρουμε ποιοι είναι οι κοινωνικά εμπλεκόμενοι και ποια θα είναι ε, τα αποτελέσματα. Γι' αυτό ο Ευρωπαίος φορολογούμενος θα πρέπει να ενημερώνεται και όχι μόνο σε κεντρικό επίπεδο στις Βρυξέλλες, αλλά και στα κράτη και περιφερειακά. Ελπίζω τα πράγματα να μην αποφασίζονται και κλεισμένων των θυρών και να μπορέσουμε να κρίνουμε καλύτερα αυτή την αξιολόγηση. Γι' αυτό είμαι σίγουρη ότι θα κάνετε τη σωστή αξιολόγηση αντικτύπου, κυρία Επίτροπε. Θέλω να είμαι σαφής. Όλοι έχετε χρονομιλίας που και η κατανομή γίνεται από τις πολιτικές ε, ομάδες. Όμως δεν είναι σωστό να διαβάζετε με τέτοια ταχύτητα. Δεν είναι σωστό για κανέναν, διότι διαβάζετε με τέτοια ταχύτητα που είναι αδύνατον να γίνει η διερμηνία. Θα ήθελα να αρκεστείτε στο χρόνο σας, αλλά να μιλάτε σχετικά αργά. Ο κύριος Μαριάς από το ECR η αξιολόγηση των ε, επιπτώσεων της νομοθεσίας της ευρωπαϊκής ένωσης είναι μια σημαντική δραστηριότητα. πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει στο πολιτικό πεδίο διότι σε πρώτη φάση οφείλει η επιτροπή να εξετάσει την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα πάρα πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με τις ίδιες τις αρμοδιότητες της ευρωπαϊκής ένωσης με την προστασία της αρχής των δωτών εξουσιών με την προστασία της τήρησης του τεκμηρίου αρμοδιότητας υπέρ των κρατών μελών. αυτό είναι το πρώτο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να εξετάζει η ευρωπαϊκή επιτροπή. το δεύτερο θέμα είναι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων διότι αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία ενέχουν πολλές προβληματικές και πολλά ζητήματα. τρίτο οι επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τέθηκε. πραγματικά πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. θα σας φέρω ένα παράδειγμα στην ελλάδα όπου εφαρμόζεται το μνημόνιο και όπου δεν έγινε καμία, κανένας έλεγχος καμία αξιολόγηση των επιπτώσεων των κοινωνικών των οικονομικών όπου έχουμε χιλιάδες ανέργους όπου έχουμε χιλιάδες φτωχοποιημένους έλληνες θα σας πω τι συνέβη κύριε επιτροπέ διότι η επιτροπή είναι και μέλος της τρόικας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 230.000 επιχειρήσεις έχουν κλείσει. Μείωση του τζίρου 75%. Φορολογικές υποχρεώσεις δεν μπορούν να εκπληρωθούν το 46% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθυστερεί τις πληρωμές. Αν είχατε κάνει μια εκτίμηση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων, πράγματι θα είχαμε ενδεχόμενα διαφορετικά αποτελέσματα. Πρέπει επίσης να έχουμε εκτίμηση των επιπτώσεων για την τεχνολογική ανάπτυξη, διότι χωρίς τεχνολογία δεν μπορούμε να περάσουμε στο νέο παραγωγικό μοντέλο. Αυτά λοιπόν πρέπει να γίνουν και σε επίπεδο Κομισιόν, βεβαίως και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Υποδειγματικό ο συνάδελφο. Ευχαριστούμε πολύ, Παύλ Φελίτσκα, για την ομάδα των φιλελευθερών. Τα τελευταία χρόνια περιμέναμε περισσότερο από το Κρήτο νομοθετή. θέλαμε λιγότερο γραφειοκρατικό φόρτο, τον αυξήσαμε. Θέλαμε απλούστερη νομοθεσία, την περιπλέξαμε. Δεν είμαστε συνεπείς και επιβαρύνουμε περισσότερο και τις επιχειρήσεις και τους πολίτες χωρίς να επιτυγχάνουμε καλύτερους στόχους. Η καλύτερη νομοθεσία είναι κορυφαία προτεραιότητα. Ε, το είπα και στο παρελθόν, και στη διοίκηση και στις επιχειρήσεις με τις οποίες συζητώ. Είναι το πρώτο, η πρώτη ή δεύτερη προτεραιότητά μας. Καλό είναι να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος κατά 10-15%. Θα είχαμε αύξηση κατά 1% του ΑΕΠ. Είναι σημαντικό θέμα, με σημαντικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Τώρα, δεν είναι θέμα μόνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βεβαίως ε, προχώρησε, μπορεί να προχωρήσει περισσότερο. Το Συμβούλιο ε, δεν έκανε τίποτε. Το Κοινοβούλιο πρέπει να προχωρήσει περισσότερο. Αυτό είναι θέμα διοργανικής συμφωνίας. Μπορεί να γίνει στο μέλλον. Πρέπει η αξιολόγηση αντικτύπου να είναι κεντρικό θέμα για την καλύτερη νομοθεσία θα έπρεπε να γίνεται ανεξάρτητη αξιολόγηση με επαγγελματισμό, ε, με ειδικού επαγγελματίες, με τη ε, μεγαλύτερη δυνατή ανεξαρτησία. Ο Αντιπρόεδρος θα πρέπει να ε, παρακολουθεί και να εποπτεύει όλα αυτά. Οι οικονομικοί στόχοι πρέπει να υπάρχουν. Είναι φιλόδοξο αυτό, αλλά λειτουργήσε και σε κάποια κράτη-μέλη και στην Αμερική. Ε, απευθύνθηκα στον Αντιπρόεδρο, θα ήθελα να κάνω κι εγώ παρόμοιε ερωτήσει όπω ο κύριο Πίπερ, δεν θα τι επαναλάβω. Η φιλοδοξία του είναι ενθαρρυντική, θέλουμε να ε, συνεργαστούμε, σίγουρα θα σα υποστηρίξουμε, αλλά θέλουμε αυτά αποτελέσματα, όχι όπω προχωρήσαμε τα προηγούμενα δέκα χρόνια. Ευχαριστώ. Επόμενο ο μιλητής, ο κύριο Ράινχαρτ Μπιούτικ για του Πρασίνους. 1,5 λεπτό. Θα προσπαθήσω σε 1,5 λεπτό να διατυπώσω τρεις απλές σκέψεις. Πρώτον, πρέπει να προσέξουμε ώστε το θεματολόγιο για την καλύτερη νομοθεσία και ρύθμιση να μην γίνει πρόσχημα για άλλο θεματολόγιο της, ε, της ε, ε, μη ρύθμισης. Βλέπω την Ευρώπη σήμερα να καταστρέφει μελλοντικές ευκαιρίες της οικονομίας μέσα από την απορρίθμιση. Είναι σημαντικό η αξιολόγηση αντικτύπου να παραμείνει ένα συνεκτικό εργαλείο για να μην αλλάξει το θεματολόγιο μας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το κόστος αλλά και τα πλεονεκτήματα των ρυθμίσεών μας, της νομοθεσίας μας. Θα πρέπει να δούμε ενδεχομένως ποιες νέες αγορές θα δημιουργηθούν. Αυτά πρέπει να τα δούμε μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Δεύτερον, η ομάδα των εμπειρογνωμόνων ε, της Επιτροπής ε, πρέπει να εργαστεί πολύ συγκεκριμένα. Τονίζω ότι οι εκπρόσωποι των καταναλωτών, των, του κλάδου της υγείας, των φορολογουμένων στην ομάδα αυτή αποστασιοποιούνται. Πρέπει λοιπόν να, συζητήσουμε προσεκτικά. Δεν θα πρέπει να ε, δημιουργήσουμε ένα γραφειοκρατικό ομολόχ ε, που θα μιλάει για την απογραφειοκρατικοποίηση και θα πρέπει να ε, βοηθήσουμε τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να εξαιρεθούν από πολλές ε, επιβαρυντικές νομοθεσίες. Ευχαριστώ ο κύριος Ντομινίκ Μαρτά, 1,5 λεπτό. Μια εγγεγραμμένη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαιρετίζουμε τη φρόνηση της Κομισιόν πριν αναλάβει οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία διότι θέλει να ζυγιάσει τα υπέρ και τα κατά των πολιτικών επιλογών που διαθέτει μέσω με ενό εξανυχιστικού ελέγχου των πιθανών αποτελεσμάτων τους. Δεν αφισβητώ την αξιοπιστία, αν και είναι πολλά τα λόμπι και αποτελεσματικά εδώ μέσα. Αναρωτιέμαι όμως για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου τελικά και το κόστος της. Μόνο όταν στριμωχτεί κανείς, όταν φτάσει και δει τον τοίχο πολύ καλά, τότε αναγνωρίζει την ικανότητα του χτίστη. Εδώ βλέπουμε ότι πεθαίνει η βιομηχανία μας, αυξάνεται ενδυμικά η ανεργία, χάνεται η αγοραστική δύναμη, αποτυγχάνουν τα συστήματα παιδείας, υπάρχει ανεξέλεγκτη εισρωή ξένων και χάνονται οι αξίες και έχω ξεχάσει πολλά. Εξηγείται σωστά ότι κάθε αξιολόγηση που βοηθάει στη λήψη αποφάσεων αλλά δεν την υποκαθιστά. Πρόκειται τελικά πάντοτε για μια πολιτική απόφαση που λαμβάνει το σώμα της Επιτροπής στο σύνολό του και το εγκρίνει, το επικυρώνει το Κοινοβούλιο. Επομένω, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, πού βρίσκεται το λάθος. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μπόνι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο για την ε, κινητοποίηση της οικονομίας καθώς και τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να βελτιώσουν την πρόσβαση σε καινούριους πελάτες αλλά η συνεχής και συνεχώς αυξανόμενη γραφειοκρατία δεν διορθώνεται μόνο από μία αξιολόγηση. Γι' αυτό χρειάζεται διαφάνεια και για τις αξιολογήσεις αντικτύπου για να εξεταστούν, να λάβουν υπόψη τους και τα πρόσθετα βάρη που φέρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις πιθανές και δυνατές επιπτώσεις που θα είχε ένα ανεξάρτητο σώμα αξιολόγησης αντικτύπου. Και τι εννοώ ανεξάρτητο, εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που να ορίζει και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν από κοινού. Μαζί πρέπει να το κάνουμε. Η Κομισιόν, τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο γιατί μπορεί να προωθήσει συνολικές λύσεις για την καλύτερη νομοθεσία και μπορεί επίσης να ενισχύσει τη μείωση του γραφειοκρατικού άκθους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε όμως τα μέσα για να το πράξουμε αυτό, να βελτιώσουμε τις συνθήκες λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την απλοποίηση της γραφειοκρατίας. Ευχαριστούμε Μάκιντάιρ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Παρακολούθησα τις παρατηρήσεις του Αντιπροέδρου της Επιτροπής η αξιολόγηση του αντικτύπου βελτιώνει την νομοθεσία και μειώνει το κόστος της νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Θέλουμε ρυθμιστικό πλαίσιο που θα προωθεί την καινοτομία, τις ειδικευμένες θέσεις εργασίας και πρώτη πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι ανάγκες όλων των επιχειρήσεων διαφοροποιούνται. Δεν είναι δηλαδή ενός μεγέθους όλες και θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε την προσέγγιση που θα τις βοηθήσει. Εμείς ως βουλευτές θα πρέπει να αξιοποιήσουμε ε, πρώτα την αξιολόγηση αντικτύπου που έχουμε στο Κοινοβούλιο και πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Θέλω να ρωτήσω την Επικομισιόν συγκεκριμένα, να ζητήσω να ε, δημοσιεύονται οι, αντίκτυποι, οι αξιολογήσεις των αντίκτυπων ε, και να προβλέπονται εξαιρέσει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Κυρία Βίξτρομ, ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, διαπιστώνουμε ότι οι προθέσεις σας ε, συμπεριλαμβάνουν καλύτερη ποιότητα των αξιολογήσεων αντικτύπου. Με αυτό συμφωνούμε και εμείς γιατί είναι σωστό να υπάρχει νομοθεσία πιο αποτελεσματική αλλά και πιο διαφανής. Είναι κάτι που θα ήταν πολύ καλό και για τους πολίτες και για ολόκληρο το Κοινοβούλιο ανεξαρτήτως πολιτικών κομμάτων. Εγώ είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών και μπορούμε και μέσω αυτής να επηρεάσουμε τη ζωή των πολιτών. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε πώς ακριβώς δουλεύουν τα πράγματα. Πρέπει επίσης να έχουμε τα μέσα που χρειάζεται η εφαρμογή της πολιτικής αυτής για μέσω μιας καλύτερης ανάλυσης των αποτελεσμάτων. Ελπίζω να μπορέσετε να τα διαχειριστείτε όλα αυτά με μεγάλη προσοχή και εγώ θα είμαι από τις ενθερμότερες υποστηρίκτριές σας αν το πετύχετε. Καπέλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, κύριε Αντιπρόεδρε, Επίτροπε Τίμερμανς, μας είπατε απόψε πόσο σημαντική είναι η αξιολόγηση αντικτύπου για την ανάπτυξη την απασχόληση στην Ευρώπη και είπατε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να βοηθήσουν να καταπολεμηθεί η απασχόληση. Συμφωνώ. Η Ευρώπη χαρακτηρίζεται από ΜΜΕ, ε, υπάρχουν ε, το 99,8% των επιχειρήσεων ε, είναι σε αυτή την κατηγορία και πάνω από 90 εκατομμύρια απασχολούμενοι είναι στις επιχειρήσεις, δηλαδή το 1 τρίτο των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα είναι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν η νομοθεσία και η αξιολόγηση που θα πρέπει να εντοπίζονται ε, στις ε, ΜΜΕ. Συμφωνώ με την πρόταση του κυρίου Πίπερ, ε, θα πρέπει αυτά τα τεστ για τις ΜΜΕ να είναι πάλι δεσμευτικά. Think small first. Αυτό πρέπει να είναι η αρχή μας για να είναι ε, φιλική η νομοθεσία μας προς τις ε, ΜΜΕ. Η κυρία Σάντερ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, τα τρία τέταρτα των ε, Ευρωπαίων κρίνουν ότι υπάρχει υπερβολική γραφειοκρατία. Κάτι το οποίο στην ουσία κατακαιρματίζει στην Ευρώπη. Οι ΜΜΕ που αποτελούν το 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι και τα πρώτα θύματα και οι μελέτες δείχνουν ότι το διοικητικό κόστος μιας νομοθεσίας είναι 10 φορές υψηλότερο για τις ΜΜΕ σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή λεπτομεριακές διαδικασίες έτσι ώστε η νομοθεσία μας να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ΜΜΕ, σε αυτή τη δοκιμή ΜΜΕ. Αυτή η δοκιμή αφορά το ίμιση των νέων κειμένων. Ακόμα χειρότερα, οι νέε κατευθυντήριε γραμμέ τη Επιτροπή για την αξιολόγηση αντικτύπου δεν κάνουν λόγο για αυτή τη διαδικασία. Ενώ γίνεται διαβούλευση για το Small Business Act και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς κινητοποιούνται για να εισακουστούν, η Επιτροπή δεν θα πρέπει να κατεβάσει τον ε, πύχη. Θα πρέπει να μας ενδιαφέρει ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, αν θέλουμε η Ευρώπη να είναι χρήσιμη και να βοηθά τις ΜΜΕ. Κάλλας, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Οι μικροεπιχειρήσεις είναι ο βασικός γνώμονας για την ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα πρέπει να μπορέσουν να ανθίσουν. Γι' αυτό θα πρέπει οι νόμοι να είναι κατάλληλοι και να ισχύουν και για τις ΜΜΕ όπως και για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, ε, το κόστος για τις ΜΜΕ είναι 10 φορές υψηλότερο για να συμμορφωθούν σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό δεν πρέπει να ισχύει. Η Επιτροπή θα πρέπει να βρεθεί στη θέση ενός μικρού επιχειρηματία, ο οποίος δεν μπορεί να συμμετέχει σε τέτοιες βαρισίμαντες διαβουλεύσεις. Ποια είναι η διαδικασία για να βοηθήσουμε τις μικρές επιχειρήσεις στα πλαίσια της μελέτης αντικτύπου. Έχετε μπλε κάρτα, τη δέχεστε, Μπόγκοβιτς. Ο κύριος Μπόγκοβιτς. Έχετε μισό λεπτό. Έχω μια ερώτηση. Ερώτηση σχόλιο. Νομίζω ότι πρέπει να ορίσουμε σαφέστερα σε ποιους τομείς θα απλουστευτούν οι διαδικασίες. Οι δημόσιες συμβάσεις είναι ένας τομέας νομίζω όπου αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ τα μεγαλύτερα προβλήματα. Είναι ένας από τους τομείς αυτός στην Ευρώπη όπου υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Συμφωνείτε μαζί μου. Όπως ξέρετε, οι μπλε κάρτες έχουν σχέση με ερωτήσεις. Εσείς τη διατυπώσατε την τελευταία στιγμή. Κυρία Κάλλας, θέλετε να απαντήσετε. Συγγνώμη, αλλά δεν άκουσα την διερμηνία, άρα δεν είμαι σε θέση να απαντήσω. Ακούγα μια άλλη γλώσσα, όχι τη δική μου. Ο κύριος Μπόγκοβιτς ε, στην ουσία προέβησε ένα σχόλιο και όχι σε ερώτηση. Γκάμπους, για μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Τίμερμαν, θα ήθελα να τονίσω τη μεγάλη σημασία για τις ΜΜΕ της σωστής μελέτης αντικτύπου του Ευρωπαϊκού Ρυθμιστικού Πλαισίου. Στην Καταλωνία εγκρίναμε πέντε νόμους τα τελευταία τρία χρόνια για να μειώσουμε την γραφειοκρατία, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ που είναι δύσκολο να προσαρμοστούν σε νέο διοικητικό φόρτο. Και μην ξεχνάτε ότι αυτές είναι που απασχολούν το 70% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτόμαστε σε μικρή ε, κλίμακα, όπως ορίζεται στο Small Business Act. Η ΜΜΕ είναι πραγματικά η ατμομηχανή της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας. Δημιουργούν πλούτο και θέσεις εργασίας. Γι' αυτό θα πρέπει ε, έτσι να προωθήσουμε την ε, πολιτική μας δράση. Θεωρούμε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να βελτιώσει αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο δεν αρκεί. Θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι και να έχουμε καλύτερες κατευθυντήριες γραμμές για την ε, βελτίωση και την αποδοτικότητα του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου για να υπάρχει ε, ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Στέφανετς, για 1,5 λεπτό επίσης. Σε πανενουσιακό επίπεδο είναι ουσιώδες να γνωρίζουμε τις επιπτώσεις των αποφάσεων που λαμβάνουμε Επομένως η ποιότητα των αξιολογήσεων αντικρύπου είναι ουσιώδης για την αξιολόγηση της λειτουργίας της Ένωσης. Τρία θέματα θέλω να θίξω. Πρώτον, πιστεύουμε ότι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Κάθε απόφαση και ψήφισμα πρέπει να βασίζεται σε αυτό το κριτήριο και προτεραιότητα. Αυτό βέβαια έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι οι μεγαλύτεροι εργοδότες. Δεύτερον, η Κομισιόν έχει ταυτίσει 10 προτεραιότητες και πρέπει να γνωρίζουμε τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτή η νομοθεσία για τον κάθε τομέα. <clears throat> Και τα, δεν πρέπει να υπάρχει επικάλυψη των κριτηρίων ή αντιφάσεις μεταξύ τους. Αντίθετα πρέπει να είναι συμπληρωματικά και να διασυνδέονται μεταξύ τους. Και τέλος, το τρίτο, θα ήθελα να τονίσω τον ουσιώδη ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως μόνο εκλεγμένο οργάνου της Ένωσης και προσβλέπω σε συνεργασία με την Κομισιόν στην αξιολογήσει της αντικτύπου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Για 1,5 λεπτό τώρα η κυρία Πάνοβα. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, συχνά σκεπτόμαστε πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον και να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι, αντιμετωπίζουν ΜΜΕ. Πρέπει λοιπόν να, να ιεραρχήσουμε τα προβλήματα για να μειώσουμε το διοικητικό φόρτο. Ε, αυτό το θέμα είναι μια προτεραιότητα της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προσπαθεί να βελτιώσει την νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχαρητήρια για την ενδιαφέρουσα ομιλία σας νωρίτερα απόψε. Think small first, να σκεφτόμαστε σε μικρή κλίμακα πρώτα. Αυτή η αρχή πρέπει να εφαρμοστεί περισσότερο. Με ε, υποχρεωτικό τεστ των ΜΜΕ για την αξιολόγηση των ε, νομοθεσιών. Οι ΜΜΕ ζουν σε συνθήκες ε, σκληρού ανταγωνισμού και η μικρότερη μείωση του διοικητικού φόρτου μπορεί να είναι πολύ σημαντική για αυτές. Ε, δεν καταλαβαίνω και δεν ε, θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός ότι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές ε, δεν αναφέρουν το τεστ των που πρέπει να θεωρηθεί υποχρεωτικό στοιχείο στη διαδικασία αξιολόγησης αντικτύπου και θα πρέπει να υπάρχει. Υπάρχει μπλε κάρτα, τη δέχεστε? Η κυρία Γκραπίνη. Όχι, δεν τη δέχομαι. Εντάξει, καλώς. Ο κύριος Λαβριέ. Ναι, ναι κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να σας πω ότι βάσει αυτών που μας είπε η Κομισιόν για τις εξολογήσεις αντικτύπου θα ήθελα να θυμίσω ποιος είναι ο αρχικός στόχος είναι ένα εργαλείο για τη νομοθετική δουλειά απαραίτητο για να γνωρίζουμε αντικειμενικότερα ποιες θα είναι οι επιπτώσεις των αποφάσεών μας που πολλές φορές δεσμεύουν τα κράτη-μέλη και επιβαρύνουν και τον πολίτη. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε πάρα πολύ οι αξιολογήσεις αυτές να μην είναι η μοναδική πηγή της νομοθεσίας ούτε τη μιας αλόγης της αύξησής της ή μείωση των της ελευθερίας του επιχειρήν. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωκομισιόν να προσέξει να μην κάνει άκαμπτες όπως ήταν μέχρι τώρα αναλύσεις και να σας δώσω και μία συμβουλή λίγο αστεία χιουμοριστική να μην χρειαστεί ποτέ αξιολόγηση αντικτύπου για τις αξιολογήσεις αντικτύπου, να μην φτάσουμε εκεί. Ωραία, τελείωσε ο κατάλογος των ομιλητών και τώρα το Catch διά η κυρία Σουίκα πρώτη. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε ότι 85% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες. Άρα είναι πολύ σημαντικές για την οικονομία. Κύριε Τίμερμαν, οι προθέσεις σας και είναι πολύ ενθαρρυντικές και είπατε ότι χρειάζεστε την υποστήριξή μας, θα την έχετε μάλλον, αλλά έχουμε και ερωτήματα και απορίες όταν δημιουργηθεί αυτό το ανεξάρτητο σώμα αξιολογήσεων που θα δώσει περισσότερο κύρος στην νομοθετική μας διαδικασία θα σημαίνει αυτό ότι η δική μας υπηρεσία αξιολογήσεων θα επικαλύπτει την άλλη. Εάν γίνουν σωστά οι αξιολογήσεις αντικτύπου, αν μειωθούν τα βάρη, αν απλοποιηθεί η νομοθεσία, και είναι εύληπτη και ευεφαρμόσιμη, γιατί να χρειάζεται αυτό το νέο ανεξάρτητο σώμα. Αυτό να μας εξηγήσετε. Ο κύριος Καπούτος. Ευχαριστώ. Η αξιολόγηση αντικτύπου έχει μεγάλη σημασία για τους πολίτες. Ε, δυστυχώς όμως έχουν διπλή όψη. Νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επίτροπη να ορίσει αυτές τις αξιολογήσεις αντικτύπου όχι με βάση πολιτικά ιδεολογήματα, αλλά με βάση καθαρά επιστημονικά δεδομένα. Θα πρέπει να βασιστούμε σε επιστημονικά καθαρά δεδομένα και να προωθήσουμε ένα νέο σύστημα συλλογής δεδομένων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε τις ε, πολιτικές μας ε, επιλογές έτσι ώστε οι αξιολογήσεις να είναι πραγματικά ε, ακέραιες και διαφανείς. Ο κύριος Πόλτσακ έχει το λόγο. Εν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, θέλω να υπογραμμίσω και εγώ ότι αυτός ο τομέας με ενδιαφέρει πολύ, γιατί είμαι νομικός και ξέρω ότι εκατομμύρια ε, πολίτες ζητούν καλή νομοθεσία. Όταν η Κομισιόν ζητεί αλλαγή της τωρινής νομοθεσίας, η πρόταση δεν ε, συνοδεύεται ε, από το μεταφρασμένο κείμενο και δεν μπορούμε να κάνουμε καλή σύγκριση μεταξύ του παλιού και νέου προτινωμένου κειμένου. Ακόμη, πρέπει να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο του κανόνα της επικουρικότητας ιδιαίτερα στα πλαίσια της ε, Λισαβόνας και των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα μπορούσατε να μας πείτε πώς θα μπορούσατε να είσαστε πιο αξιόπιστοι στις αξιολογήσεις αντικτύπου. Γιατί τις περισσότερες φορές ε, πρόκειται για μια τυπική διαδικασία που υπηρετεί τα μεγάλα ευρωπαϊκά λόμπι. Εσείς όμως δυστυχώς δεν δίνετε καμία αξιοπιστία σε αυτό το μέσον. Δήθεν κινείστε υπέρ των ΜΜΕ. Θέλετε να διευκολύνετε τη ζωή των ΜΜΕ τη στιγμή που κατατροπώνονται στην εσωτερική αγορά. Όπως συνέβη στην Πορτογαλία με την παρέμβαση της Τρόικας. Επίσης ε, υπηρετείτε τις περισσότερες φορές τους μεγάλους ε, ομίλους και εκείνο κοινοπραξίες και γι' αυτό οι ΜΜΕ έπρεπε στην ουσία να υπηρετήσουν τα ολιγοπόλια και τα μονοπόλια ε, του τομέα των τηλεπικοινωνιών και ούτω καθεξής. Ο κύριος Τίμερμανς έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου για τους διερμηνείς, διότι οι ομιλητές μιλάνε τόσο γρήγορα που έχω εντυπωσιαστεί από τη δουλειά των διερμηνέων. Δεύτερον, ας λύσω μια παρεξήγηση. Η αξιολόγηση αντικτύπου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι τμήμα των σχεδίων μας και θα παρα... ήταν παρέμ και θα παραμείνει. Το μόνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε τις διαδικασίες. Να σας πω πώς δουλεύει η υπηρεσία της Επιτροπής που προετοιμάζουν την νομοθεσία και αυτές την χάνουν αξιολόγησης που την εξετάζει το αρμόδιο όργανο και δυστυχώς μέχρι τώρα πολλές φορές μας έλεγαν ότι δεν ήταν καλή η αξιολόγηση. Πρέπει λοιπόν οι ίδιες μας οι υπηρεσίες να δουλεύουν καλύτερα κατά την αξιολόγηση αντικτύπου. Και αυτό που κάνουμε τώρα είναι να αναθεωρούμε τις κατευθυντήριες γραμμές για να δουλεύουμε καλύτερα. Και αυτά που είπατε σήμερα είναι για μένα πολύτιμα για να διασφαλίσω την δημιουργία καλύτερων κατευθυντηρίων γραμμών. Η υπόθεση ότι οι αντιξιολογήσεις αντικτύπου δεν θα γίνουν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα περίπου 93% των προτάσεων έχουν αξιολογήσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, νομίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε και τη λειτουργία του οργάνου αξιολόγησης, διασφαλίζοντας ότι του Συμβουλίου, αν θέλετε, αξιολόγηση, διασφαλίζοντας ότι τα μέλη του θα είναι πεπειραμένα, σαφώς ανεξάρτητα και θα μπορούν να πούν και με βίο ακόμη τρόπο αν χρειάζεται στην Κομισιόν ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Έχω την πρόθεση να εξετάσω πολύ καλά τη σύνθεση του. Μερικοί πρότειναν να μην είναι τμήμα της ε Κομισιόν. Αυτό, με αυτό διαφωνώ νομίζω. Πρέπει να παραμείνει μέρος της Κομισιόν, αλλά να γίνεται η αξιολόγηση πριν έρθουν τα κείμενά μας, τα, οι προτάσεις μας στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Και θα συνεννοηθούμε και με το Κοινοβούλιο, θα δούμε πώς κάνει εκείνο τις αξιολογήσεις του και μήπως και εμπνευστούμε. Η αξιολόγηση αντικτύπου σημαίνει εξέταση του αντικτύπου στην ευρύτερη κοινωνία, όχι μόνο της νομοθεσίας όχι μόνο είναι καλογραμμένη η νομοθεσία, αλλά ποιε είναι οι οικονομικές της, ποιος είναι ο οικονομικός της αντίκτυπος, ποιος είναι ο περιβαλλοντολογικός τη αντίκτυπο. και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την καλύτερη νομοθεσία. Η κυρία Ταντίτσκα είπε ότι θα έπρεπε ίσως να έχουμε και δημοσιονομικούς στόχους για την καλύτερη νομοθεσία. Λοιπόν, Νομίζω ότι και ο κύριος Μπουτικόφερ το είπε. Καλύτερη νομοθεσία δεν σημαίνει απορρίθμιση αναγκαστικά, ούτε η λιγότερη νομοθεσία. Μπορεί να σημαίνει η αντικατάσταση 28 εθνικών νομοθετημάτων από ένα ενωσιακό, αλλά μπορεί επίσης να σημαίνει ότι η Ένωση δεν νομοθετεί σε ορισμένα θέματα, γιατί ο αντίκτυπος θα ήταν τόσο τεράστιος ώστε θα μπορούσε να επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για μένα που το βλέπω λογικά δεν είναι ιδεολογικό θέμα και πολιτικά αντικό, είναι θέμα λογικής. Πώς θα εξασφαλίσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη χωρίς να επιβαρύνουμε ιδιαίτερα τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αυτός είναι ο στόχος τα επόμενα πέντε χρόνια. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε την υπάρχουσα νομοθεσία. Δεν το έχουμε κάνει αυτό. Η κυρία Ταντίτσκα νομίζω σωστά το έθιξε αυτό. Και θέλω διάλογο με το Κοινοβούλιο για να δούμε και πώς θα μπορούσαμε να αφαιρέσουμε παροχημένη νομοθεσία ή νομοθεσία που δεν επιτυχάνει τους στόχους που ήθελε να πετύχει. φυσικά επειδή υπάρχουν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά επίσης και επειδή η υποβοήθησή τους θα ήταν ευκολότερο να έχει μεγάλο αντίκτυπο από ότι να επηρεάσουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις θα ήταν σωστό να τονίσουμε ιδιαίτερα τη σημασία τους για να έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα αλλά έχω την εντύπωση ότι μέχρι τώρα ό,τι και να κάναμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν το αίσθημα ότι τους αφαιρούμε βάρη αλλά μερικές ότι τους προσθέτουμε. Ότι το μόνο που κάνει η Ευρώπη είναι να προσθέτει βάρη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και να κάνουμε κάτι απτό και συγκεκριμένο για αυτές. Αποκινούμε την και με το Κοινοβούλιο. Και για να συνοψίσω κυρία Πρόεδρε, μάλιστα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα παραμείνουν τμήμα των αξιολογήσεών μας, θα είναι καλύτερες οι αξιολογήσεις από ό,τι τα τελευταία ένα-δύο χρόνια και αυτό είναι τμήμα της καλύτερης νομοθεσίας που είναι απαραίτητη. Και επίσης, ναι, η Κομισιόν αναλαμβάνει τη δέσμευση όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να παίξουν πλήρως το ρόλο που πρέπει να παίξουν και ελπίζω αυτό να το δείτε και στις καινούργιες διευθυντήριες γραμμές που θα σας υποβάλουμε σύντομα. Ευχαριστούμε κύριε πίτροπε. Λίγη η συζήτηση και θα ψηφίσουμε την Πέμπτη. Περνάμε στο τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι οι παρεμβάσεις διαρκείας ενός λεπτού. Θα αρχίσουμε με τον κύριο Χέις για ένα λεπτό. Μικρόφωνο.